Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας για αυτή τη Σύνοδο Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια συζήτηση που ήταν ε, πιο ε, φορτισμένη από ό,τι συνήθως ε, γιατί ξέρουμε ότι την Πέμπτη το μεσημέρι πολλές φορές οι συζητήσεις είναι πολύ βαρετές αλλά τώρα ήταν πολύ